ζήτησε το, να πάρει το λόγο εξ ονόματο του Συμβουλίου ο υπουργό Λοπέ Γαρίδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Χαίρομαι που δίνετε την ευκαιρία να παρέμβω και σε αυτό το σημείο τη διάταξη, το οποίο αφορά την κοινωνία των πολιτών αλλά και τις μειονότητες στην Λευκορωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα προβληματίζεται πολύ όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης στην Λευκορωσία. Ειδικότερα δε μας προβληματίζουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φήμωση της ελευθερίας του λόγου, η αύξηση της ε, καταστολής της βάρος των ΜΜΕ. Νόμοι, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση του διαδικτύου. Πράξεις κατά της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων της. Όλα αυτά είναι μια επιδείνωση της ε, κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Is την δήλωση της 16ης Δευτέρα η κυρία Άστον τοποθετήθηκε και επίσης εξέφρασε ανησυχία για τα όσα γίνονται εις βάρος της πολωνικής μειοψηφίας στην ε, Λευκορωσία για τις ε, φυλακίσεις κάποιων μελών της κοινότητας της πολωνικής στις οποίες προέβη η αστυνομία και αυτού του είδους η επίσημη δήλωση και θέση της υψηλής εκπροσώπου διαβιβάστηκε στις ε, λευκορωσικές αρχές μέσω των διπλωματικών εκπροσώπων τους. Τη Δευτέρα συζητήθηκε στο Συμβουλίο των και εμβαθύναμε σε αυτό το θέμα. Θα επαναληφθεί αυτή η συζήτηση και έλαβε το λόγο ο Πολωνός υπουργό, ο οποίος επίσης εξέφρασε ανησυχία. Επίσης εξέφρασε την αντίθεσή του και το ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε κατά αυτής της συστηματικής δίωξης της ε, πολωνικής μειονότητας. Επίσης θα πρέπει να σας αναφέρουμε ότι Οπότε, όλος ο κόσμος μπορεί να πούμε με λίγα λόγια ότι παρακολουθεί την κατάσταση με ανησυχία και προβληματισμό και από κοντά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει το μήνυμα στις λεωφορικές αρχές ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους δεσμεύσεις. Στον ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προστασία των μειονοτήτων. Μια από αυτά είναι ε, σημαντικό τμήμα της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων, αλλά και στο Συμβούλιο Εξωτερικών είπαμε ότι ερητά ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους Υπουργούς ούτως ώστε από τους κατάλληλους διάβλους και όπου είναι σωστό να επισύρουν την προσοχή των όσων συμβαίνουν υπό πλευράς των αρχών της Λευκορωσίας. Θα πρέπει επομένω να καταφέρουμε με πίεση να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα και για να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τα δικαιώματα αυτή τη μειοψηφία στη Λευκορωσία που παραβιάζονται και ταυτόχρονα. Είναι σημαντικό η Λευκορωσία να προχωρήσει προς την σωστή κατεύθυνση. σοβαρά τις σχέσεις μας μαζί της και στα πλαίσια των πολυμερών διεθνών της σχέσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δήλωση της ε, Προεδρίας ε, του Συμβουλίου αναφέρθηκε στις θέσεις της ΥΠΑ του εκπροσώπου της Βαρόνης ε, Άστον που έχει εκφραστεί πολύ έντονα για το θέμα αυτό. Θα ήθελα πάνω σε αυτά να προσθέσω δύο λόγια για την ισχυτική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, ιδίω σε σχέση με την πολωνική μειοψηφία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα οπισθοχώρησης ε, των προσπαθειών για τον εκδημοκρασμό της Λευκορωσίας τα τελευταία χρόνια του τελευταίου, θα πρέπει να παραμείνουμε σε διάλογο με τη Λευκορωσία, να αφήσουμε ανοιχτές τι διάβλους επικοινωνίες όσο δύσκολο και αν είναι. Και αυτό όχι μόνο με τα ε, επίπεδα της ε, κυβέρνησης, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και επαφές ε, σε ατομική βάση που είναι πάρα πολύ σημαντικά παραδείγματος χάρη με ανταλλαγές φοιτητών με ευκαιρίες επιχειρησιακές πολιτιστικές αναλλαγές ε, σαν ε, μια πλατφόρμα επικοινωνίας με τους πολίτες της Λευκορωσίας σαν μια δυνατότητα για να διατηρήσουμε τη δυνατότητα πρόθεσης της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Και τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι παρόλη την αντιστροφή της κατάστασης τα δύο τελευταία χρόνια, η Κομισιόν θα ήθελε να παραμένει δεσμευμένη εκεί και να συνεχίσει να ακολουθεί μια επιτάχυση θετικής διαδικασίας. για να ξαναβρεθούμε στην κατάσταση που είμαστε πριν από δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ των ε, των πολιτικών ομάδων τώρα, ο κύριος Χόκμαρ, καταρχήν για τη δική του ομάδα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ισπανική Προεδρία και την Επιτροπή για τα όσα είπαν για την κατάσταση. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε σαφείς ε, σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό για το οποίο συζητάμε ε, γεγονός είναι οι ενέργειες μιας δικτατορίας και ενός βίου καθεστώτος που αρνείται τα δικαιώματα των μειονοτήτων καθώς και τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα στη Λευκορωσία και αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο κίνησης πιστεύω για τις συζητήσεις μας για τον διάλογο με το καθεστώς. Ένα διάλογος, ο διάλογος μάλλον θα πρέπει να είναι αμφίδρομος. Και όταν θα ξεκινήσει ο διάλογος θα πρέπει να απαιτήσουμε από το καθεστώς της Λευκορεσίας, μάλλον απαιτήσαμε να αλλάξουν, να κάνουμε τα ρυθμίσεις, να προχωρήσουν σε αλλαγές τις οποίες δεν έκαναν. Και θα πρέπει να υπογραμμίσω εντόνως ότι δεν είναι πολωνικό ζήτημα. Η Λευκορωσία είναι στην γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβάνεται στην ανατολική εταιρική σχέση. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και με τις δράσεις μας τώρα, τις ενέργειές μας τώρα, το καθεστώς της Λευκορωσίας, μάλλον τις δράσεις του, με τις δράσεις του το καθεστώς Λευκορωσίας απομακρύνεται και απομονώνεται από μόνο του ε, και απομακρύνεται και από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα πρέπει Κάθεται να ζητήσουμε σεβασμό μειονοτήτων μειονοτήτων, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πάυση των βιωτήτων της αστυνομία και προθυμία για επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω πως το μήνυμα αυτό θα πρέπει να είναι ε, ξεκάθαρο προς το καθεστώς. Ο διάλογος μας θα πρέπει να είναι ένας διάλογος για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βεβαίως θα πρέπει να στραφούμε στην κοινωνία των πολιτών Γιατί η Λευκορωσία είναι πολύ περισσότερα από το καθεστώ. Είναι ο κόσμος που ζει εκεί. Φοιτητέ, άνδρες, γυναίκες, η κοινωνία. Και πιστεύω ότι αυτό που είδαμε τελευταία απέδειξαν ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε σε διάλογο άμεσα με την κοινωνία των πολιτών για να ενισχύσουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία και τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κρίστιαν Βίγενίν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εξ ονόματο τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θα ήθελα να εκφράσω τι ανησυχίε μα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και ιδιαίτερα όσον αφορά τι πρόσφατε εξελίξει ε, για την Ένωση των ε, Πολωνών. Ε, θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα με του πολίτε τη Λευκορωσία που δεν είναι σε θέση να χαίρουν των βασικών του πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο γεγονός και όλοι συμφωνούμε από αυτό. Και αυτό είναι και το σημείο κίνηση. Και η κύρια ερώτηση που πρέπει τώρα να θέσουμε είναι καταρχήν πότε πού θέλουμε να φτάσει η Λευκορωσία και δεύτερον πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Για το πρώτο νομίζω συμφωνούμε όλοι. Θέλουμε η Λευκορωσία να είναι, γίνει δημοκρατική, οι αρχές της Λευκορωσίας δημοκρατικά να, εκλεχθούν, να εκλεγούν, δηλαδή το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος, οι τοπικοί α, εκπρόσωποι, να υπάρχει μια ελεύθερη ατμόσφαιρα και βεβαίω η χώρα να κινηθεί πιο κοντά προς την Ένωση. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει την πολιτική της προς τη Λευκορωσία από την απομόνωση στην επαφή. Και φαίνεται πως αυτή η πολιτική δίνει κάποια αποτελέσματα. Βέβαια αυτό δεν αρκεί, δεν γίνεται αρκετά γρήγορα και οι εξελίξεις που βλέπουμε στα τελευταίες ε, δύο εβδομάδες δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε πιο προσιλωμένοι στο θέμα. Ε, θα μεταβούμε με την αποστολή ε, μας στην Λευκορωσία να δούμε την κατάσταση επιτόπου και έχουμε μια κοινή στρατηγική με τα τρία όργανα, Συμβούλιο, Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Χρειάζεται μια τέτοια στρατηγική για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αλλήλων και να δημιουργήσουμε το πολιτικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη πολύ συγκεκριμένο για τη Λευκορωσία, όχι μόνο γενικέ συστάσεις, αλλά ένα πρόγραμμα δράση το οποίο θα πρέπει να τηρήσει η Λευκορωσία. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Δεν είναι αρκεί να γίνει μόνο μέσω της οικονομική συνεργασίας υπό την ανατολική εταιρική σχέση. Σα ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματο των ε, φιλελευθέρων ο κύριος Γκερμπράντι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω πως ε, η σημερινή συζήτηση είναι μια περιφερειακή συζήτηση. Είδαμε ότι ο Γιάννου Κόβιτς εξελέγει στην Ουκρανία ένας πρόεδρος που σαφώς είναι προσανατολισμένος περισσότερο προς τη Μόσχα από ό,τι προς τις Βρυξέλλες και είναι καλό ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της επίσκεψής του δεν αφήσαμε να μας ρίξει στάχτη στα μάτια για τη Λευκορωσία. Ο, αυτά που κάνει ο Λουκασέγκο προς την πολωνική μειονότητα είναι ένα σημάδι ότι και αυτός είναι στραμμένος προς τη Ρωσία περισσότερο, προς τη Μόσχα παρά προς την ε, Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να απειμείνουμε ώστε να πάψει η μεταχείριση αυτή της ε, μειονότητας αυτής. Και αυτό όμως συμβαίνει ότι είμαστε, γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα νότα μας τραμμένα προς την ε, Ανατολή. Ανοίγουμε τα μάτια μας που και που, αλλά όχι πραγματικά προς τις χώρες αυτές. Στεκόμαστε και κρίνουμε με αυστηρότητα τα όσα κάνει η Λευκορωσία απέναντι στην ε, πολωνική μειονότητα, αλλά από την άλλη πλευρά και εμείς πρέπει να ανοίξουμε περισσότερο, να έχουμε μια πολιτική θεωρία θεωρήσεων λιγότερο περιοριστική, να εξετάσουμε τα θέματα της ενεργειακής πολιτικής. Να προσπαθήσουμε δηλαδή και να στραφούμε περισσότερο προς χώρες ε, όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία και θα πρέπει να προσανατολίσουμε το όραμά μας προς αυτές τις χώρες ώστε να έχουμε πιο θετικό αντίκτυπο σε σχέση με τις εσωτερικές εξελίξεις και όχι μόνο να παριστάνουμε τους ε, αφιψηλού δικαστές και να αφήνουμε τη Ρωσία να κάνει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουτελ, εξ των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Γιατί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι σαφές. Οι διαδηλώσεις στις οποίες συνελήφθησαν 40 Πολωνοί. Αυτό πρέπει να το κατηγορήσουμε. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό άλλο θέμα που ανέφερε και ο συνάδελφος Βικενίν. Το Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό αποφάσισε το Μίνσκ να τύχει επίσκεψη μια αντιπροσωπεία. Εγώ είμαι ένα από εκείνου του ε, τέσσερι συναδέλφου που θέλουν να πάνε εκεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια εικόνα τη κατάσταση γιατί υπάρχουν προβλήματα με την ελεύθερη έκφραση, το δικαίωμα του... Ε, κλπ. Ε, πρέπει να δυναμώσουμε, να εμβαθύνουμε τη σχέση μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη απόφαση αποτελεί επίση απόφαση. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Λευκορωσία θα, τον Μάρτιο θα χρειάζεται, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερο σήμερα. Η αντιμετώπιση των Πολωνών στη Λευκορωσία δεν είναι απλά πολωνικό ζήτημα, όπως ήδη υπόθηκε. Είναι η έκφραση μιας προσέγγισης ε, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα στάνταρ και συμπεριλαμβανομένων των ε, δικαιωμάτων των ε, μειονοτήτων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει την τήρηση των βασικών αρχών δικαίου όπως τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αν ο κύριο Λουκασέγκο δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα των ανθρωπίνων αξιών, σίγουρα καταλαβαίνει τη γλώσσα των κυρώσεων. Δεν θέλουμε κυρώσει που θα πλήξουν την ε, κοινωνία τη Λευκορωσίας, αλλά και κυρώσει που θα κάνουν τη ζωή δύσκολη στους ε, υπαλλήλου και του πολιτικού που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Έχουμε μια δυσανάλογη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει την πόρτα. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα όμω, ε, σε αντάλλαγμα. Είναι πλέον η ώρα για πολιτικέ κυρώσει να αποκλειστούν οι εκπρόσωποι των Λευκορώσων ε, στην ε, ε, διακοινοβουλευτική συνέλευση και να επανεγκαθιδρυθεί ο μαύρος, η μαύρη λίστα. Δύο λεπτά κυρία Κίνγκαγκάλ, ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι συμπρόεδρος της ομάδας ενδιαφέροντων για μειονότητες και μειονοτικές γλώσσες, οπότε δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε απόλυτα αυτά τα οποία κάνουν η Λευκορώση κατά αυτή της μεγάλης ε, οργάνωσης ε, της μειονότητας και της μειονότητας γενικότερα. Ξέρετε, κυρίως είναι ηλικιωμένοι αυτοί που το εφίστανται αυτά και τελικά ε, εδώ έχουμε παραβίαση και δικαιωμάτων μειονοτήτων και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπότε θα πρέπει όλοι εμείς που έχουμε γίνει μάρτυρες κομμουνιστικού καθεστώτος να αναγνωρίσουμε τα κοινά σημεία των όσων κάνουν σήμερα η Λευκορώση με αυτά. Οπότε γι' αυτό και όλα αυτά τα έχουμε καταγγείλει και έχουμε πει ότι είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε τέτοιο ε, οποιαδήποτε τέτοια πολιτική που εργάζεται τα δικαιώματα και είπαμε ότι θα πρέπει η υπατή εκπρόσωπος να κάνει διαβήματα προς την λευκορωσική κυβέρνηση σβαστούν τις υποσχέσεις τους, ότι θα πρέπει επίσης να, να τους πούμε ότι θα υπάρξει πάγωμα στη σχέση της χώρας με την ΕΕ. Και τα ίδια δεσμενότητα στην ανθρώπινα δικαιώματα και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί θέμα εσωτερικό ενός κράτους. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επίσης ε, θέμα πολωνολευκορωσικό ή είναι θέμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, άλλωστε είναι και θέμα της πολιτικής μας προς ε, Ανατολά, της πολιτικής γειτονίας. Οπότε θα πρέπει η Επιτροπή να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να αναλάβει και διαβήματα επίσης ξεκάθαρα. Σας ευχαριστούμε και τώρα ο 1,5 λεπτό ο κύριος Λιμπεράτσικη Εγώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω Συμβούλιο και Κομισιόν, διότι ήταν ταχεία η αντίδραση. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση πώς θα πρέπει να αντιδρούμε, αλλά ξέρετε σε αυτή την περίπτωση δεν είναι θέμα προστρεβής μεταξύ των δύο χωρών, είναι καταστολή δικαιώματος ε, ελεύθερης έκφρασης, δικαιωμάτων ανθρωπίνων, δικαιωμάτων μειονοτήτων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί και σε οποιαδήποτε άλλη μειονότητα. Τώρα μιλάμε για την πολωνική μειονότητα απλά γιατί είναι πολύ πολωνική σε μειονότητα, είναι οργανωμένη, είναι δημοκρατική και έχουν και τον Μενικέβιτς ε, εν μέσω αυτών ο οποίος έχει βραβευτεί με το βραβείο Ζαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να γιατί μας απασχολεί το θέμα τώρα. Τι να κάνουμε. Μίλησα με αυτούς τους ανθρώπους, εκπροσώπους της μειονότητας, ε, δύο φορές ήρθα στις και μου είπαν ότι δεν θέλουν οικονομικές κυρώσεις. Είναι συνεπείς πολίτες της Λευκορωσίας. Θέλουν πολιτική καταδίκη, θέλουν να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Λευκορωσίας και ΕΕ. Θέλουν να υπάρξει συνεργασία που όμως να εξαρτάται από τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Να τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει επομένω να έχουμε τέτοια αποστολή διακρύβωση ε, που θα πρέπει να πάει εκεί, να μα υποβάλει μια έκθεση και να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ένα λεπτό, κύριο Σιβάνσκε. Η συνθήκη τη Λισαβόνα, πρόεδρε, αποτελεί μια υπόσχεση για πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Όμω, ήμασταν αόρατοι στην IT. Τίποτα απλώ τα λένε τα συνεργά μεταξύ του και δεν κάνουμε τίποτα προ τα έξω. Να σήμερα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δυστυχώ αποφάσισε το Συμβούλιο να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων. Το ΔΕ Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, έστω και έχουμε τόσο κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων. Και πρόκειται για χώρα τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Επίτροπε, απέτυχε η πολιτική των ανοιχτών θυρών σταματήστε αυτές τις ανταλλαγές των φοιτητών και σπουδαστών που μετά από μία πενταετία έχουν καταστρέψει την αξιοπιστία μας και έχουμε γίνει ένας κομπάρ στη διεθνή σκηνή και το ξέρει αυτό και η Μόσχα και η Ουάσιγκτον. Να σταματήσουμε αυτές τις θολές αντιδράσεις. Ε, dziękuję panie przewodniczący. Ε, jako szef delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią το θέμα των ε, σχέσεων με την ε, Λευκορωσία είναι ένα θέμα το οποίο ε, μας προκαλεί διαρκώς πρόβλημα. Ακούω τα διάφορα επιχειρήματα που λένε ότι η Λευκορωσία έχει δικαίωμα στο δικό της ρυθμό για να εκδημοκρατιστεί και να φτάσει στα ε, ισχύοντα στάνταρ. Ε, θεωρητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ασκήσει πίεση επί κυρίαρχων χωρών ε, αν λάβαμε υπόψη την, όσον αφορά την εσωτερική της κατάσταση. Με αυτό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αν δεν υπήρχαν και διεθνείς προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται και η Λευκορωσία θα πρέπει να τα δεχτεί σε ένα μικρό μέρος ε, στο κέντρο της Λευκορωσίας πρόσφατα οι αρχές καταχράστηκαν ε, τη ε, ισχύω των αστυνομικών έναντι μιας ομάδας ηλικιωμένων συνταξιούχων που είχαν συγκεντρωθεί με δική τους πρωτοβουλία και θέλανε να μετατρέψουν ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης σε ένα κέντρο ε, των ε, πολωνικής κουλτούρας. Και τι έκανε το καθεστώς. Έστειλε την αστυνομία. Αρχικά δεν άκουσε καν τους μάρτυρες ενώπιον ε, του δικαστηρίου για να αποδείξει το τι έκαναν ε, ήταν δικαιολογημένο. Και να, όταν γίνεται κάτι τέτοιο δεν, γίνεται, δεν υπάρχει σεβασμός για τα διεθνή στάνταρα. Η Λευκορωσία είχε όμως ε, δεχτεί να τα τηρήσει όταν ξεκίνησε τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανατολική εταιρική σχέση, η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να συνδέεται με την εγκατάλειψη τέτοιου είδου πρακτικών και μια πραγματική απελευθέρωση και εκδημοκρατισμό τη χώρα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλές ε, παρεξηγήσεις για, ε, για την πολωνική μειονότητα στην Λευκορωσία που θα πρέπει να επιληχθούν χωρίς ε, βία. Εγώ θέλω να υποστηρίξω την θέση της Επιτρόπου για τη συνέχιση της ε, συνεργασίας και της επαφές σε ανθρώπινο επίπεδο. Αύριο η πρώτη αντιπροσωπεία θα πάει στην Λευκορωσία. Προσβλέπουμε σε ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο με τις αρχές. Θα επιστρέψουμε με τα συμπεράσματα μας και ίσως θα έχουμε και προτάσεις της Λευκορωσίας για την συμμετοχή στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις μας. Και η, Λιδία θα είναι οι τοπικές ε, εκλογές ε, στις 25 Απριλίου. Θα πρέπει να υπάρχει εκεί ε, μια πραγματική εκλογή και να μην ακολουθήσουν όλοι την ίδια γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες επίνεσε την Ένωση για την ταχεία αντίδραση. Όμως, χάρη στην πολιτική του ομάδα, σήμερα δεν προβαίνουμε σε έγκριση ψηφίσματος. Κάθε μέρα δουλεύει η Επιτροπή στα θέματα της ανάπτυξη και αν σήμερα έρθει και μας πει κάποιε προτάσεις, μα ποιος θα είναι χαρούμενος. Αν μας τα πει αυτά η, η Επίτροπος που βλέπει εξελίξεις και η ίδια που από τα πέντε λεπτά που μίλησε αφιερώνει δύο σε αυτό το θέμα. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει την ευκαιρία μας δόθηκε για να τοποθετηθείτε. Εμείς έχουμε πει ότι απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο το οποίο προσφέρεται τόσο ώστε να προσθέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μιλάμε τώρα για πολωνούς, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Μπάουρε να μισή λεπτό. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι η Λευκορωσία καταπιέζει την πολωνική μειονότητα. Φυλακίσεις, εκφοβισμοί και είναι δηλαδή τελικά μια πάγια τακτική της Λευκορωσίας. Εγώ προέρχομαι από την Σλοβακία και εγώ είμαι μέλο μια μειονότητας και καταλαβαίνω τι τραβάνε η Πολωνία εκεί. Αυτά τα οποία καταγγέλει η κυρία Μπορή ε, από την Λευκορωσία. Γιατί πολλέ φορές η συμπεριφορά προ μια μειονότητα είναι σαν να πρόκειται για έναν εχθρό για κάποιον αλυτρωτιστή οπότε είναι όλα αρνητικά έχουμε τέτοιους παρενόχληση πίεση είναι πάει στα αυτές αδεσμοί δημοκρατικών καθεστώτων. Να δούμε όμω υπόψη ότι τα δικαιώματα τη μειονότητα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το βεβαιώνει ο ΙΕ. Επομένω, έχουμε τώρα διακρίσει, διακρίσεις, έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων, ε, τέτοιου είδους ε, εκφοβισμό. Όλα αυτά δεν μπορεί να θεωρούνται εσωτερικό θέμα μια χώρα. Είναι απαράδεκτα. πρόκειται για εκβιασμό, πρόκειται για απειλές. Αυτά δέχονται και οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου που πάνε στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει επομένω και εμεί να στείλουμε ένα μήνυμα στην Λευκορωσία ότι δηλαδή μια τέτοια πολιτική σοπαίδευση των μειονοτήτων είναι κάτι το απαράδεκτο. Και τώρα κάτσε τη Πρόεδρο. Ένα λεπτό. Μίκλος. τόση ώρα ακούω με προσοχή τα όσα μας ε, αναπτύσσει η κυρία Επίτροπος. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα να είναι πιο δυναμική η αντίδρασή της. Αυτά που λέτε σήμερα από τα πριν δύο εβδομάδες όταν γίνανε όλα αυτά τα γεγονότα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να λάβουμε δράση. Σήμερα κάποιοι μιλούν για κυρώσεις. Μα ήδη έχουμε αποφασίσει για κάποιες κυρώσεις, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Λέμε για υποστήριξη των πολιτών, αλλά όποιος πήγε εκεί πέρα, είδε ότι βρίσκεται, είναι τη γενέστηση η κοινωνία των πολιτών εκεί. Άρα να κάτσουμε και να σκεφτούμε ότι κάθε χώρα έχει κάποιες υποχρεώσεις έναντι των πολιτών. Και να δούμε πώς θα στηρίξουμε κάποια ανεξάρτητα ΜΜΕ που υπάρχουν στην χώρα εκείνη. Και τηλεόραση ανεξάρτητα. Και να δούμε πώς θα δώσουμε ευκαιρίες σε φοιτητές από τη χώρα εκείνη να έρθουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, λέει το μικρόφωνο σας, το τον επόμενο ομιλητή, Κύριε Νίτρας. Κυρίε και κύριοι, στην προηγούμενη θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε διάφορα ψηφίσματα για τη Λευκορωσία όταν ε, καλούσε το καθεστώς να σταματήσει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την καλή της βούληση και δεν χρησιμοποίησε κυρώσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη επιθετική πολιτική ε, του λευκορωσικού καθεστώτος απέναντι στις μειονότητες, ιδιαίτερα την Πολωνίκη, είναι πολύ ανησυχητική με ένα έτος πριν από τις εκλογές. Οι, πολιτικές, οι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 ε, κατάσχονται χωρίς προειδοποίηση, γίνεται εκφοβισμός των ανθρώπων ε, συμπεριλαμβανομένου του ε, νικητή του βραβείου Ζαχάροφ θα πρέπει να ψηφίσουμε ένα κατάλληλο ψήφισμα αλλά και να καλέσουμε τις αρχές της Λευκορωσίας να κάνουν κάτι πια και επίσης η κυρία Άστον με βάση το άρθρο 33 της συνθήκης θα πρέπει να συστήσει την θέση του ειδικού εκπροσώπου που παρακολουθεί την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή σχόλιο. Ο κύριος Λίσεκ, ένα λεπτό. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι είναι καλό που αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα της Ρευκορωσίας εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά δεν αρκεί βέβαια να μιλάμε. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσουν να συνεχίσουν ένα στρατηγικό σχέδιο που θα ε, μας πει πώς θα υποστηρίξουμε τις μη κυβερνικές ε, οργανώσεις και τα ελεύθερα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση στην ε, Λευκορωσία. Συζητάμε για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά ε, πράγματα που είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα, αλλά αδιαφέροντα, αλλά αυτονόητα για μας και εκείνους είναι όνειρο μόνο. Περιμένουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να βρει ένα στρατηγικό σύστημα για να βοηθήσουμε την κοινωνία εκεί. Κύριος Λίσεξ, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ο πρόεδρος θα δώσει το λόγο στον κύριο Λόπες Καρίζο. Ευχαριστώ. Μετά από όλα όσα ακούσαμε δεν μπορώ εγώ παρά να συμφωνήσω. Να συμφωνήσω με όσα καταγγέλουν οι βουλευτές για τις παραβιάσεις των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Διότι Φύγεται εν προκειμένου η πολωνική μειονότητα. Α, επομένως φύγεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο γιατί πρόκειται για μειονότητα προσώπων που σχετίζονται εθνοτικά με κράτος μέλος Ένωσης. Όμως, πρόκειται για σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων μειονότητα. Επομένως και άλλες καταγωγές να ήταν αυτή η μειονότητα, πάλι θα ήταν το θέμα σοβαρό. Μια που πρόκειται για δικαιώματα παγκόσμιου χαρακτήρα εδώ που θυγόνται. Γι' αυτό επομένω αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λέγαμε τα ίδια, ακόμα και αν πρόκειται για άλλη μειονότητα. Είναι αδιαίρετα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι παγκόσμιο χαρακτήρα. Οφείλω να σας πω ότι το ότι έχουμε από ένα καθεστώ τέτοιες παραδιάσεις αυτό δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να ζημιωθούν οι πολίτες της χώρας αυτής. Φυσικά είναι σημαντικό το ότι έχουμε εδώ πέρα κάποια χώρα που συμμετέχει στην, ε, ε, στην πολιτική μας ε, για, την πολιτική γετνίαση, το people to people και άρα θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επαφή, ξεκάθαρη, άμεση, που να αφορά τη δική μας επικριτική στάση σε σχέση με αυτές τις παραβιάσεις. Αυτό που το κάνει η κυρία Από κοντά παρακολουθεί εξελίξεις, όπως και ο πρόεδρος Μπούζεκ, που έρχεται κιόλας σήμερα, τώρα στην έδρα. Θα πάει σε αμέσως μέρες στο Κίεβο η κυρία Άστον ε, για την, ε, για την έλευση των ε, καθηκόντων του κυρίου Κέβιτς. Εκεί θα πάει στον κύριο Λουκασέγκο, οπότε βεβαίως και πρόκειται και να ενεργήσει αναλόγως προς αυτόν. Όλα αυτά θα προσκόψουν και το Συμβούλιο Εξωτερικών της Ένωσης. Μια που είναι θέμα μεγάλη σημασίας. Και γι' αυτό και είναι θετικό το ότι σήμερα συζητήσαμε στον Ολομέλεια το θέμα αυτό ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και τώρα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Γεωργίευα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Καταρχήν να ευχαριστήσω για τη συζήτηση σε αυτή την αίθουσα και να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο για, τον, για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί και το θεμέλιο επί του οποίου η σχέση με οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένης της Λευκορωσίας στηρίζεται και η, ο παραβίαση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία είχε έφτασε σε ένα ατυχώ ε, ε, σκοτεινό και χαμηλό σημείο πρόσφατα, αλλά δεν ξεκίνησε με αυτό. Ξεκίνησε από τις αρχές του 2009, πράγμα το οποίο οδήγησε τον Νοέμβριο του 2009 το, το Συμβούλιο Υπουργών να ζητήσουν από την Κομισιόν να διατυπώσει πρόταση για την, το αποκαλούμενο κοινό ενδιάμεσο πρόγραμμα για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από την Λευκορωσία. Οι υπηρεσίε τη Κομισιόν προετοίμασαν ένα σχέδιο αυτού του ενδιάμεσου προγράμματο για τι μεταρρυθμίσει. Τώρα είναι στα χέρια του είπα εκπροσώπου που της είπα εκπροσώπου που θα δεχτεί και τα πορίσματα της αποστολής έρευνας που στέλνει εκεί το Κοινοβούλιο αύριο. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, Ε, θα, ληφθεί, θα, θα σχηματιστεί ε, το τελικό πρόγραμμα δράσης και μεταρρύθμισης. Το δεύτερο ήμιση του 80, της δεκαετίας του 80, ξεκίνησε η Περιστρόικα στην πρώην Σοβιετική Ένωση και οδήγησε σε, ε, για πρώτη φορά για τη ζωή πολλών σε μια ευκαιρία να υπάρξουν ε, ανταλλαγές ε, φοιτητών και, φοιτητών και καθηγητών, ε, εμένα συμπεριλαμβανομένης και με οδήγησε στη London School of Economics. Σίγουρα μου άλλαξε τη ζωή και βοήθησε να βοηθήσω με τη σειρά μου τη χώρα μου. Και γι' αυτό τον ανοίγουμε τα δημοκρατικά κανάλια, τους διάβλους για χώρες υπό καταπιστικά καθεστώτα, γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα και να επαναλάβω την παρατήρησή μου για τη σημασία και τη χρησιμότητα των ανθρώπινων επαφών, της χρησιμότητας της στήριξης των επιχειρήσεων, της διατήρησης των επαφών παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τα πολύ σοβαρά προβλήματα των μειονοτήτων τα οποία καταδικάζουμε. Επαναλαμβάνω, ζητώ να μείνουμε σε επαφή ε, έτσι ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τον λαό της Λευκορωσίας ώστε να, προχωρήσουν, να προχωρήσει σε ένα δρόμο ελευθερίας και σύνδεσης με την Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, που αφορά το Πεκίνο 15 χρόνια μετά προφορική ερώτηση της κυρίας Εύα